Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε στις θέσεις μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε τις εργασίες της υποεπιτροπής μας. Ε, το θέμα μας ε, σήμερα, μάλλον τα δύο θέματά μας, είναι δύο εκθέσεις, ε, όπως καθορίσαμε εδώ. Η πρώτη έκθεση είναι Πασκού ρήτρε αμοιβαία άμυνα και ελεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση του κύριου Πασκού. Το λόγο έχει ο κύριο Πασκού, γιατί θα έχουμε τεράστιο όγκο στοιχείων ε, για τη συζήτηση και μετά από την ε, Θεσμική Επιτροπή, επειδή έχουμε πετύχει μια συμφωνία και ευχαριστούμε τον Άντριου. Με την Επιτροπή την ΕΦΚΟ έχουμε πετύχει μια συμφωνία, άρα λοιπόν θα συνεργαστούμε στενά με εκείνους για τη θεσμική πτυχή ακριβώς, για το τι γίνεται, πώς αυτές οι δύο ρήτρε που συμπεριλαμβάνονται στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ε, τι γίνεται με αυτές. Κύριος Πασκού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν δύο, κάνα δύο πράγματα που πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι η γενική εικόνα είναι ότι το Συμβούλιο πρέπει να επεξεργαστεί μια απόφαση προς το τέλος του χρόνου αυτού. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ακουστεί έγκαιρα η φωνή του Κοινοβουλίου, ώστε να επηρεάσει το Κοινοβούλιο την απόφαση αυτή. Τώρα, η έγκριση της έκθεσης προβλέπεται για το, τη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου. Οπότε θα υπάρχει χρόνος αρκετός, νομίζω, για να μπουν σωστά κάποια πράγματα εγκαίρως. Τώρα, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος, η ΑΦΚΟ μέσω του ε, συναδέλφου μας ΔΑΦ έχει κοινή ευθύνη για θεσμικά θέματα με βάση τον κανόνα 50. Ο κύριος ΔΑΦ είναι εδώ και θα πει και εκείνο τη γνώμη του στη συζήτηση αυτή και είναι ευπρόσδεκτη γνώμη του στην έκθεσή μας. Τώρα υπάρχει μια γενικότερη στρατηγική εικόνα εδώ. Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με όλο και πιο κοντινούς, κοντινές απειλές που προσεγγίζουν τα σύνορά μας. Παράλληλα, εμείς όλο και περισσότερο γινόμαστε έσωστρεφείς και αφιερώνουμε όλο και λιγότερους πόρους για την άμυνα και την ασφάλειά μας. Και το πρόβλημα της προστασίας των πολιτών μας καθίσταται αναπόφευκτο, αν και μπορεί να μην θέλουμε να το αναγνωρίσουμε ως υπάρχουν πρόβλημα τώρα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι κανένα κράτος μέλος της Ένωσης δεν μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει τις όλο και πιο περίπλοκες απειλές για την ασφάλεια. Η αλληλεγγύη είναι κέρια και αυτό είναι ένα κομμάτι της εξίσωσης. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να αναγκάσουμε και να πιέσουμε τα κράτη να ξεπεράσουν αυτό που θεωρούν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια πολύ λεπτή ισορροπία εδώ μεταξύ αλληλεγγύης και αρκετή ελευθερία στα κράτη-μέλη από την άλλη για να επιλέγουν αν θα στηρίξουν κάποιο κράτος μέλος και πώς. Αυτό, αυτές οι δύο ρήτρε υπάρχουν εδώ και τρία χρόνια στη συνθήκη της Λισαβόνας και δεν έχουμε κάνει πολλά για να δούμε πώς σε περίπτωση που ένα κράτος ζητήσει ενεργοποίηση της ρήτρα, αυτή θα γίνει. Ελπίζω αυτό προς το τέλος του χρόνου να αποσαφινιστεί. Δεν ζητάμε να δημιουργηθούν άλλα μέσα και μηχανισμοί. Αυτό που κάναμε με τις συζητήσει με τον κόσμο στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο ήταν να κάνουμε μία απογραφή των υπαρχόντων μέσων για να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και να συναρμολογούνται αν θέλετε και να συνεργάζονται για να έχουμε ε, επαρκή απόκριση σε μια τέτοια περίπτωση. Κάναμε μια συζήτηση για τη ρήτρα της ε, αμοιβαίας άμυνας ε, που την πήραμε από τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, ένας όρος που επίσης χρησιμοποιείται. Μάλιστα προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε όλα αυτά με μία ε, υποσημείωση στην έκθεση, γιατί η αλλαγή του τίτλου της έκθεσης τώρα συνεπάγεται πολλή γραφειοκρατία και πολλά πράγματα που μπορεί να μας εκτροχιάσουν από το στόχο μας που είναι να είμαστε στην ώρα μας για τη συζήτηση στο Συμβούλιο στο τέλος αυτού του χρόνου. Η σχέση με το ΝΑΤΟ είναι σημαντική, διότι 21 χώρες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή καλύπτονται από τη συνθήκη του ΝΑΤΟ και υπάρχει ε, άμεση μνήα αυτού. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν καλύπτονται και θα πρέπει να επαφίενται σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που θα χρειαστούν την υποστήριξή μας. Και εδώ όντως πρέπει να δούμε σοβαρά τη σχέση αυτή με τη συμμαχία. Παράλληλα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που υφίστανται και στους δύο οργανισμούς και παράλληλα θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις εδώ. Σε ό,τι αφορά τις δομές και τις διαδικασίες, καλούμε την ύπατη εκπρόσωπο να προτείνει πρακτικές διευθετήσεις σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος θελήσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα μηδέας συνδρομής υπάρχει και θέμα ενός επιχειρησιακού κέντρου της Ένωσης που είναι από πολιτική άποψη πολύ λεπτό θέμα. Νομίζω ότι ξέρετε ότι αναπόφευκτα ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το εξετάσει κάποια στιγμή αυτό πολύ σοβαρά. όμω, πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή προς αυτή, προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι γνωρίζετε πάντως ότι αυτό θα καταστεί αναπόφευκτο στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αλληλεγγύης, η έκθεση είναι αρκετά λεπτομερής εδώ. Ακόμα και αν θέλαμε δεν θα αποφεύγαμε κάποιες τεχνικές πτυχές. Νομίζω ότι ξέρετε ότι η βασική αρχή εδώ είναι ότι η ρήτρα αλληλεγγύης θα πρέπει να την πρέπει να την επικαλούνται κράτη όταν είναι σαφέστατο ότι ξεπερνούν, η κατάσταση ξεπερνά τις ικανότητές τους, με άλλα λόγια δηλαδή δεν ε, είναι μια επιχειρησιακή, ένα επιχειρησιακό αίτημα που θα το υποβάλει ανά πάσα στιγμή μια χώρα, όποτε θέλει. Πρόκειται για σοβαρή απόφαση όταν ε, αποφασίσει την ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας ένα κράτος μέλος. Στο παρόν πλαίσιο της οικονομικής κρίσης είναι ε, σημαντικό τα κράτη-μέλη να εντοπίζουν λύσεις ε, για την κοινή ανάπτυξη στην περίπτωση ε, όπου οι πόροι είναι υψηλού κόστους. Κάποιες χώρες που έχουν τέτοιους πόρους καμιά φορά είναι απρόθυμοι να διαθέσουν τους πόρους αυτούς σε άλλους. Παράλληλα όμως, αν χρειαζόμαστε αυτή του, ε, ε, αυτούς τους ειδικού πόρους και διατυπωθεί το σχετικό αίτημα, θα πρέπει να βρούμε μία ε, λύση μέσα από το λεγόμενο pooling and sharing, δηλαδή τη συνένωση και κοινή χρήση των πόρων στην άμυνα και την ασφάλεια, που θα πρέπει να ισχύει η συνένωση των πόρων και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το τομέα. Σε ό,τι αφορά τη συνοχή της δράσης, αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί αυτό που θέλουμε είναι μια ταχεία απόκριση αντίδραση σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ε, σε αυτή την περίπτωση η ταχεία απόκριση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις εισρωές από όλους τους φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ούτω ώστε να υπάρξει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εάν εγώ περιμένω από κάποιον να δώσει τη συμβολή του στη διαδικασία και καθυστερήσει αυτός ο κάποιος, ο κάποιος φορέας, τότε η κατάσταση επιτόπου θα επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν μια άλλη ισορροπία που πρέπει να βρεθεί. Σίγουρα υπάρχουν αναπόφευκτες γραφειοκρατίες που θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και θα πρέπει να βρούμε Ε, ευέλικτες φόρμουλες που θα επιτρέπουν συνεργασία και να μην υπάρχει κάποια ερμηνεία, δηλαδή ότι κάποιος μπαίνει στα χωράφια άλλων. Η ιδέα είναι όλοι να συμβάλλουν στην επίλυση κάποιου συγκεκριμένου προβλήματος που θα αναφύεται. Υπάρχει εμπειρία δεδομένη, επί της οποίας μπορούμε να στηριχτούμε και η οποία υπάρχει και στο επίπεδο του Συμβουλίου αλλά και κυρίως στο επίπεδο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτή η εμπειρία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί τα καλά θα πρέπει να τα διατηρήσουμε και τα υπόλοιπα να τα βελτιώσουμε. Αυτά και τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ιδιαίτερα ρεαλιστική η αντιμετώπιση. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό που είναι πολύ ευαίσθητος. Ο κύριος Ντεφ ε, από την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Πασκού διότι το σχέδιο έκθεσης είναι πάρα πολύ καλό, σόφρον, πάνω σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα. Είναι ιδιαίτερα καλό το σχέδιο έκθεσης εις ό,τι αφορά την αξιοποίηση και τους τρόπους εφαρμογής της ρήτρα αλληλεγγύης που τα παρουσιάζει με μεγάλη λεπτομέρεια. Και αυτό είναι απαραίτητο. Και ε, ως ε, πρότυπο για μας στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να μάθουμε και να εκτιμούμε περισσότερο αυτά που ήδη υπάρχουν και έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Εστιάζω λοιπόν πρώτα στο άρθρο 42 σημείο 7 που προτιμάει να το λέει ρήτρα μηδέας ε, άμυνας ε, το κ. Πασκού. Εγώ προτιμώ τη ρήτρα μηδέας συνδρομής γιατί εν μέρη γιατί 22 από τους 28 καλύπτονται εις ό,τι αφορά την αμοιβαία άμυνα από το ΝΑΤΟ. Θα ήταν λοιπόν σωστό ως Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρρύψουμε ένα ταμπού από το παρελθόν το οποίο μας έκανε να ντρεπόμαστε να μιλάμε για τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πραγματικά ένα έκτακτο γεγονός ότι ε, έχουμε την έδρα μας στην ίδια πόλη, αλλά σπάνια ερχόμαστε σε επαφή και μιλάμε ο ένας με τον άλλον ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, είναι ένα πρόβλημα το οποίο με δεξιότητα και ένα ε, βαθμό θάρρους μπορούμε να ξεπεράσουμε. Βέβαια, βέβαια ο κύριος Πασκού έχει δίκιο όταν λέει ότι κάποια κράτη-μέλη δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ για διάφορους και ειδικού ιστορικούς λόγους που δεν είναι πάντα ίδιοι και έχουν περάσει εδώ και καιρό οι εποχές κατά τις οποίες μπορούσαμε να περιγράψουμε τα κράτη μη μέλη του ΝΑΤΟ ως ουδέτερα κράτη. όπως συνηθίζαμε να αποκαλούμε τις χώρες αυτές ε, την εποχή του ψυχρού πολέμου. Όλες απολάβουν και θα συνεχίσουν να απολάβουν την, ε, της ε, ασπίδας ασφαλείας του ΝΑΤΟ, είτε θέλουν είτε όχι. Και δεν υπάρχει τρόπος ενεργοποίησης του 42-7 αν δεν υπήρχε στενή συνεργασία και επαφή με το ΝΑΤΟ. Και είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ένα σενάριο, μια περίπτωση, μια περίσταση όπου αν μια περιφέρεια της Ένωσης θα υφίστατο επίθεση θα αρνεί το να συμμετάσχει το ΝΑΤΟ. Το μόνο πιθανό σενάριο είναι μια νέα έκρηξη της ε, κρίσης μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Και ανοίγω μια παρένθεση για να απευθύνω έκκληση στο Κοινοβούλιο να είναι πολύ πιο ε, δραστήριο προβλέποντας μελλοντικές εξελίξεις. Ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών ε, και να απαγώσουν τις ε, συγκρούσεις. Εμείς ε, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε περισσότερο από ό,τι καταφέραμε στο παρελθόν. Και αναφέρομαι εδώ στην κάθε Άστον με την ιδιότητά της ως είπα της εκπροσώπου. Τώρα, δεύτερο επίπεδο σχέσεων ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι πιστό αντίγραφο των καθηκόντων του Πίτερσμπεργκ που αναφέρονται στο άρθρο 43 τώρα της συνθήκης της Λισαβόνας και δεν πρέπει να αυτά πατώμεθα ότι δεν προσπαθούν οι δύο οργανισμοί να δημιουργήσουν διευθετήσεις προς την ίδια κατεύθυνση για να κάνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτό γίνεται με πολύ στενότερη... Χρειάζεται όμως ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ μας. Σε λειτουργικό επίπεδο η συνεργασία νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακή αν και διακριτική και όχι πολύ διαφανής. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο υπολείπεται. Δεν έχει αναπτυχθεί όπως πρέπει. Πρότεινα λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και η ύπατη εκπρόσωπος να αναζητήσουν επισήμως να δημιουργήσουν, να εγκαθιδρύσουν μια ε, πολιτική συνεργασία τακτική. Πάμε τώρα στο άρθρο 222. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ θα ήθελε να υπογραμμίσει Κάποιος μου παίζει μουσική. Θέλει λοιπόν η ΑΦΚΟ Επιτροπή να πει ότι η απόφαση του Συμβουλίου έχει δύο μέρη. Το μη στρατιωτικό και το στρατιωτικό σκέλος, δύο σκέλη έχει. Και είναι σημαντικό το Συμβούλιο να καταλάβει ότι η, η ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να ισχύει ως μέθοδος ψηφοφορίας για μη στρατιωτικά χαρακτηριστικά της απόφασης. Αυτό θα διευκολυνθεί αν η ΚΟΠΣ και ΚΟΖΗ, οι δύο επιτροπές δηλαδή που χειρίζονται την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια ε, κατέληγαν σε κοινή γνωμοδότηση επί του σχεδίου απόφασης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Κομισιόν. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε σαφώς ότι δεν πρόκειται μόνο για το άρθρο 222, το οποίο αναφέρει την έννοια της αμοιβαίας αλληλεγγύης σε περίπτωση κρίσης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά έχουμε και το 122 άρθρο, το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί σε κάποιες περιστάσεις για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν κρίσεις. Και το άρθρο 196 που είναι η ρήτρα για την πολιτική προστασία. Θα πρέπει τα τρία αυτά άρθρα να τα δούμε ως ένα ενιαίο σύνολο νομικών βάσεων, αν θέλετε. Αυτά τα τρία δημιουργούν μια ενιαία νομική βάση για την εφαρμογή των διευθετήσεων που θα απαιτηθούν σε ώρα κρίσεων. Τέλος, για την προσέγγιση της ΑΦΚΟ. Νομίζω ότι είμαστε προκατηλημένοι κατά της δημιουργίας νέων θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Εκτός ε, αν πρόκειται για μια συνέλευση που θα τα προσεγγίσει πιο σοβαρά. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα για υπέρ ενός επιχειρησιακού κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικός μου πρόεδρος της ε, ομάδας Άλντε είναι ιδιαίτερα υπέρ αυτής της ιδέας, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι αν γίνει, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ πιο προσεκτικά το θέμα πριν αποφασίσουμε να το βάλουμε σε εφαρμογή και να, δημιουργήσουμε το επιχειρησιακό κέντρο. κυρία Γιαννάκο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Πασκού για την έκθεσή του η οποία επισημαίνει και όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το να δημιουργηθεί μία ρήτρα αλληλεγγύης για την άμυνα και την ασφάλεια αλλά και ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα μπροστά λαμβάνοντας υπόψη και την εργασία που έχει γίνει μέχρι σήμερα σας θυμίζω ότι από το 2003 υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις. Ε, και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει δικούς της μηχανισμούς οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με τη συμμετοχή των περισσότερων χωρών σε άλλους οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζω κύριε Πρόεδρε ότι η Ένωση αποκτά με τη συνθήκη της Λισαβόνας ενιαία νομική προσωπικότητα και ένας οργανισμός που έχει ενιαία νομική προσωπικότητα μπορεί να κάνει τα πάντα. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αναστέλει τη δυνατότητα της Ένωσης και να ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και να δημιουργήσει μια κοινή πολιτική άμυνας την οποία άλλωστε προβλέπει σαφέστατα το άρθρο 42. Το άρθρο 42 της συνθήκης μιλάει για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Τα σημειώνω αυτά γιατί είχαμε χθε μια συζήτηση στην ε, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και δεν νομίζω ότι το συμπέρασμα που βγήκε θέλω να πω στον κύριο Νταφ είναι ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συμφωνεί μαζί του ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν συμφωνεί πρώτον με την διαγραφή της έννοιας της ρήτρας άμυνας όπως θέλει να το διαγράψει ο κύριος Νταφ και δεύτερον η, Ευρω... η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Ε, αναφέρθηκε επίσης ο κύριος Νταφ στο που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια σύγκρουση. Καταρχήν τα τελευταία χρόνια μας έχουν αποδείξει ότι οι πιθανότητες δεν είναι αυτές που νομίζαμε, αλλά είναι λίγο διαφορετικές. Αλλά όντως η πιθανότητα στην οποία αναφέρθηκε έχει σημασία. Είναι δηλαδή όχι οι διαφορές μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, αλλά οι απειλές της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου. Ε, Κύριε συνάδελφοι, θέλω να σημειώσω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές Δηλαδή, τι περισσότερο μπορεί να κάνει η Τουρκία όταν δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος και ταυτόχρονα θέλει να γίνει μέλος της Ένωσης. Τι περισσότερο μπορεί να κάνει από τις γελιότητες, επιστρέψτε μου να πω, που έκανε και κάνει επί Κυπριακής Προεδρίας. Εάν η θεωρία μας είναι γενική, ότι όπου υπάρχει σύγκρουση φταίνε και οι δύο και ας το δούμε γενικώ και αορίστος και να παρέμβει το ΝΑΤΟ, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όμως, όταν οι αρχηγοί κρατών δημιούργησαν τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και όταν εμείς δουλέψαμε για την ε, ε, Ευρωπαϊκή Συνέλευση, είχαμε άλλη άποψη για, την, ε, για τη ρήτρα αλληλεγγύης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Και αυτή έχει εκφραστεί ρητός μέσα στη συνθήκη. Με όλο το σεβασμό λοιπόν στην βρετανική προσέγγιση των πραγμάτων έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη μέσω της συνθήκης αλλά και μέσω των προτάσεων του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να εξετάζουμε επί της ουσίας θέματα κοινή προσέγγισης. Και επειδή ε, σημειώθηκε και το κόστος πολύ σωστά από τον κύριο Πασκού, θα σας πω ότι παραδείγματο χάρη στο χώρο της Ευρώπης σε 16 γραμμές παράγονται τάγκς και στις Ηνωμένε Πολιτείε παράγονται σε μία γραμμή. Πληρώνουμε πολύ λιγότερα για τη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά η αποτελεσματικότητά μας είναι ελάχιστη. Δηλαδή δεν συνάδει ούτε με τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε. Επομένως είναι και δικαίωμα και υποχρέωση της Ένωσης να προχωρήσει και στον αμυντικό τομέα χωρίς αυτό να βλάψει σε τίποτα τη σχέση με το ΝΑΤΟ. Άλλωστε το να συνεργάζεται η ύπατη εκπρόσωπος με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ δεδομένο. Δεν το θεωρώ ως κάτι καινούριο. Είναι πάρα πολύ λογικό. Διότι ουδής αποποιείται τις ευθύνες του έναντι της συμμαχίας. Ούτε θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργήσει τη συμμαχία. Θέλει όμως συμπληρωματικά να βρει τρόπους να ενισχύσει την ασφάλεια των κατοίκων της Ευρώπης και αν θέλετε να ενισχύσει και την ειρήνη στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες μέσω των οποίων, με τις οποίες συνεργάζεται ε, σε επίπεδο καλής γειτονίας. Ε, άρα ε, εμείς συμφωνούμε με τον κύριο Πασκού, κάποιες τροπολογίες θα κάνουμε αλλά συμφωνούμε με την ουσία της εκθεσής του και διαφωνούμε με την προσέγγιση που κάνει ο κύριος Ντάφ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ για την έκθεση πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η έκθεση είναι πολύ συνεκτική. Όμως υπάρχουν ακόμα ασάφειες όταν πρόκειται για την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης. Νομίζω ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε πρώτον μεταξύ εδαφικής άμυνας στους κόλπους της Ένωσης και την ΚΕΠΑ για τη διαχείριση κρίσεων που είναι εξωτερική πολιτική. Το θέμα αφορά τις ικανότητες. Εμείς εννοούμε εδώ ότι χρειάζονται νέες στρατιωτικές ικανότητες να αναπτυχθούν. Τι είδους ικανότητες είναι αυτές για τις οποίες μιλάμε στα πλαίσια της ρήτρα αλληλεγγύης. Και ε, κάποια πράγματα έχουν και πολιτικές και επιχειρησιακές διαστάσεις. Βέβαια, προφανώς δεν είναι όλες οι χώρες μας ε, μέλη του ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, ε, που δεν δεν θα έπρεπε τα μη μέλη του ΝΑΤΟ να ε, συνδέονται με τα πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ και τα όπλα μαζικής καταστροφής. Επίσης, οι μάχημες ομάδες, τα battle groups θα χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσουν κομμάτι της ρήτρας αλληλεγγύης. Uh, thank you very Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο συνάδελφος Ανδρέας Νταφ εκτός από το, ότι εάν η ρήτρα αυτή αμοιβαία άμυνας όπως λέγεται γίνει τελικά αμοιβαία βοήθειας τότε ταυτίζεται πια με τη ρήτρα αλληλεγγύης και άρα μπορεί να διαγραφεί. Αυτό βασικά είπατε και συμφωνώ φυσικά με αυτό. Υπάρχουν όμως δύο χωριστά θέματα που συζητούμε εδώ και πολλοί θα συγχαίουν. Η ρήτρα αλληλεγγύη στο 222 είναι πολύ σημαντική ρήτρα και σημαίνει αμοιβαία αφημένη αλληλοβοήθεια σε περιόδους δυσκολιών και καταστροφών βασικά θα έχει μη στρατιωτικό χαρακτήρα, αλλά θα υπάρχει και κάποιο βέβαια στρατιωτική πτυχή αναπόφευκτα. Αλλά βασικά το 222 είναι ανταπόκριση πολιτικής βοήθειας, όχι στρατιωτικής. Τώρα, αυτό δεν είναι το ίδιο με το άρθρο 42, το οποίο κατ' εμένα είναι τελείως ανόητο. Όλοι οι ομιλητές μίλησαν άμεσα ή έμεσα για τον ΝΑΤΟ. Αν είστε όμως Φιλανδός ή Σουηδός και νομίζετε ότι απειλείται η χώρα σας, Πιστεύετε ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες θα σας βοηθήσει ή αν είστε και Εσθονός ακόμη ή Βούλγαρος ή Πολωνός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας βοηθήσει φυσικά όχι, το ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια οργάνωση που φέρει όλη την ευθύνη για την ασφάλεια των χωρών μας και αυτή είναι το ΝΑΤΟ. Ένα συνάδελφος μίλησε για το κόστος. Ναι, πάντα έλεγα ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα αφού γίνονται περικοπές στους ε, προϋπολογισμούς της άμυνας να δημιουργήσουμε νέα αμυντική δομή δεν μπορούμε. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι τελείως υπερβολικό για την Ένωση να θεωρεί ότι έχει δυνατότητα αμοιβαία άμυνα πέρα από εκείνη που της χορηγεί το ΝΑΤΟ. Πρέπει λοιπόν να τα χωρίσουμε τα δύο θέματα. Τουλάχιστον να υπάρχει κάποια ενθάρρυνση στο κείμενο για χώρες σαν τη Σουηδία και τη Φιλανδία ώστε να πλησιάσουν το ΝΑΤΟ και αυτές έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις της συμμαχίας ακόμη και αν δεν είναι μέλη ακόμη και αν είναι αδέσμευτες χώρες έχουν συμμετάσχει και έχουν συζητήσει με τον ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να μην επισημοποιήσουν ή θεσμοποιήσουν τη σχέση τους αυτή με τον ΝΑΤΟ. Τώρα για το Κυπριακό έχει γίνει φραγμός για πολλά πράγματα και καιρός είναι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλει να κάνει κάτι χρήσιμο να λύσει το Κυπριακό οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι δεν έχει νόημα να περιορίζονται στην περιγραφή μονόπλευρη μάλιστα του προβλήματος, το οποίο είναι πολύ πιο πολύπλοκο και υπάρχουν ευθύνες και από τις δύο πλευρές. Αν νομίσει κανείς ότι μπορεί η πλειοψηφία των πολιτών της Ένωσης να στηρίξει τους Ελληνοκύπριους για να αντιμετωπίσουν τον δίθεν τρομερό τουρκικό κίνδυνο που τους επιλεί, νομίζω ότι γελιέται όποιος το νομίζει αυτό. Πολλοί λένε βέβαια ότι δεν θα έπρεπε να ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ένωση μέχρι να λύσει το πρόβλημα με τους γειτονές της. Αυτό ήταν άλλωστε και ένα από τα κριτήρια για την ένταξη. Αλλά φαίνεται ότι το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόστηκε για την Κύπρο και αποδείχτηκε ανοιχτή πληγή από τότε. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα και γρήγορα. Αν υπήρχαν άνθρωποι καλής θέλησης και από τις δύο πλευρές και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, τότε θα μπορούσε να λυθεί. Πρέπει όμως να επιμείνει περισσότερο η Ένωση. Και τέλος Πρόεδρε, όλοι ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό πρέπει να έχουμε το πολιτικό θάρρος να προκαλέσουμε να αμφισβητήσουμε το δόγμα της Ένωσης εφόσον είναι λαθεμένο. Και όταν μιλάμε με αυτόν τον τρόπο για αυτή τη ρήτρα αμοιβαία άμυνα στη συνθήκη Λισαβόνα, δεν το πράττουμε. Ευχαριστώ. Εντάξει, έτσι ολοκληρώνουμε με το σκιοδησηγητή και τα όσα μας, θα, μας είπε ο κ. Βανόρντεν θα προκαλέσουν ορισμένες απορίες και θα δούμε, θα δούμε και για την Τουρκία και πρώτα απ' όλα όμως ε, να δούμε τις αντιδράσεις για την έκθεση αυτή, αυτή από πλευράς ε, ε, Γκουε, κ. Λίζου. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, στη γλώσσα μου μιλάμε για ρήτρα αλληλεγγύης, αυτό αφορά τις εσωτερικές πτυχές της Ένωσης και η ρήτρα της συνδρομής αφορά εξωτερικές απειλές. Και νομίζω ότι από συνταγματικής άποψης πρέπει να γίνει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των δύο, αν και υπάρχουν και κοινά σημεία. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η θέση της Γκουε ε, επιμένει στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και αυτό ισχύει και για την περίπτωση της Κύπρου. Νομίζω ότι οι Κύπροι δεν θεωρούν ότι τα προβλήματά τους θα έπρεπε να λυθούν με στρατιωτικά μέσα αλλά εμείς πιστεύουμε ότι με ειρηνικά μέσα ε, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις και με μεγαλύτερη ε, συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έκθεση την απορρίπτουμε για πολλούς βασικούς λόγους, στους οποίους δεν θα υπησέλθω λεπτομερώς, θα αναφερθώ σε ορισμένα μόνο. Ένας λόγος είναι ότι εδώ η διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται και εδραιώνεται ως μια στρατιωτική συμμαχία. Ο κύριος Στάνοκ σε μία από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΝΤΕ το είπε αυτό, το απέσυρε όμως ως λάψους λίγου, και είπε ότι είναι λάθος και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτική συμμαχία με την έννοια ε, και για την προετοιμασία αυτής της συνεδρίασης ε, μίλησα, έβαλα στο ίντερνετ τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή και βγήκε από το ίντερνετ ε, στρατιωτική συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο θέλουμε να γίνει έκθεση μειοψηφίας. Τονίζω επίσης ότι είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι η υποχρέωση αμοιβαίας συνδρομής εδώ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται με πολύ πιο αυστηρό τρόπο από ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, στο άρθρο 5 ε, του ΝΑΤΟ αφήνει ανοιχτό το ποια μορφή θα υποστηριχθεί από το ΝΑΤΟ μια χώρα που ε, υφίστανται επίθεση εδώ, βλέπουμε το στρατιωτικό σκέλος ε, να παρουσιάζεται με πιο πολλές λεπτομέρειες. Και ίσως ό,τι αφορά τις δύο ρήτρε, λοιπόν, και τη ρήτρα αλληλεγγύης, προβλήματα εσωτερικά δηλαδή, και τη ρήτρα συνδρομής, και ίσως ό,τι αφορά τις δύο ρήτρε δεν ορίζουμε τι είναι αυτό το οποίο απειλείται στρατιωτικά και όταν πρόκειται για το εξωτερικό και το εσωτερικό της Ένωσης. Ποια είναι η στρατιωτική απειλή. Είναι ας πούμε μια κυβερνοεπίθεση, είναι τρομοκρατικό πλήγμα. Τι απειλές είναι αυτές κατά των κρατών μελών της Ένωσης που θα δραστηριοποιήσουν τη ρήτρα μηδέας συνδρομής. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό ότι δεν υπάρχει ορισμός εδώ. Το ίδιο ισχύει για την υποχρέωση συνδρομής στα πλαίσια της ρήτρα αλληλεγγύης. Τι είναι καταστροφή στο εσωτερικό της Ένωσης. Και εδώ δίνω δίκιο τον προηγούμενο μιλητή, γιατί προκειμένου περί φυσικών καταστροφών ή ε, ανθρωπιστικών ε, καταστροφών θα πρέπει να σκεφτούμε την πολιτική προστασία και να δούμε με ποια μέσα θα διατεθεί η πολιτική προστασία. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε τι εννοούμε όταν πρόκειται για, ανθρωπογεν... για... για τέτοιες απειλές οι ανθρωπογενείς καταστροφές μπορεί να είναι και γενικές απεργίες. Μπορεί να είναι διαμαρτυρίες του πληθυσμού κατά της πολιτικής λιτότητας για παράδειγμα και παρόμοια. Εδώ δηλαδή θα πρέπει να το δούμε συνταγματικά το θέμα. Η στρατιωτική, ε, θα πρόκειται για στρατιωτική επέμβαση στο εσωτερικό της Ένωσης, όπως και αλλού πρόκειται για στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Αυτό σε εθνικό επίπεδο το απορρίπτουμε και βέβαια σε ό,τι αφορά το διεθνές κίνημα ε, και πρέπει να τονίσω εδώ ότι και το διεθνές κίνημα ειρήνης θα απορρίπτει όλα αυτά. Αυτό αρκεί λοιπόν για να καταλάβετε ότι από τη δική μας τη σκοπιά, από σκοπιά Γκουε και από τη σκοπιά του διεθνούς ε, φιλιρινικού κινήματος απορρίπτουμε τον βασικό προσανατολισμό της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ε, πολύ καλά και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σοφοκλέους και μετά η κυρία Γιαννάκου. Καταρχάς να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή τον κύριο Πάσκο που πραγματικά έκανε μια πάρα πολύ σημαντική εργασία και αναφίβολα πρέπει όλοι να στηρίξουμε την ενδυνάμωση αυτής της προσπάθειας ούτως ώστε η άμυνα η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ισχυροποιηθεί με ένα συγκεκριμένο και πρακτικό τρόπο και να μην περιορίζεται, θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθε, μόνο στην αλληλεγγύη που είναι χρήσιμη και στις ανθρωπιστικές ενέργειες. Όμως είμαι υποχρεωμένο παράλληλα ταυτόχρονα και λυπάμαι που θα το κάνω πραγματικά να απαντήσω στον συνάδελφο μου, τον κύριο Πανόρτη, ο οποίος άνοιξε ένα κεφάλαιο το οποίο θα έλεγα ίσως και άκερο στην Επιτροπή μας. Πρώτον, ανέδειξε ίσες ευθύνες σε μας, δηλαδή στους Ελληνοκυπρίους και στην Τουρκία. Δηλαδή έστειλε ένα μήνυμα περίπου ότι το θύμα και ο θήτης, δηλαδή ο κατοχικός στρατός, η εισβολή και η κατοχή, είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που την βιώνει για σχεδόν 40 χρόνια. Το θεωρώ πολιτικά προκλητική τοποθέτηση και απαράδεκτη τοποθέτηση. Και το δεύτερο το οποίο νιώθω την ανάγκη να υπογραμμίσω είναι ότι επίσης ανεδείχθη, επίσης άκερα, αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα δήθεν ότι υπάρχει εκείνη η σχολή που κάποιοι επέμεναν ή ίσως επιμένουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έπρεπε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθόν διάστημα δεν είχε επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εσείς το λέτε. Εμεί λέμε ότι η κυπριακή δημοκρατία έχει ενταχθεί με την προοπτική και την προσδοκία μάλιστα προσθέτω σε αυτό το σώμα ότι μαζί μας θα έχουμε συναδέρφους τουρκοκύπριους στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μία όμως προϋπόθεση ότι θα είναι λυμένο το κυπριακό πρόβλημα και περιμένουμε. Και το τρίτο που πρέπει να υπογραμμίσω και να κλείσω και το τρίτο που εδώ θα συμφωνήσω είναι ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ συμφωνώ απόλυτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικουρικό ρόλο και λόγο αλλά πρέπει να ενισχύσει την προσπάθεια. Το ερώτημα είναι προς ποιαν κατεύθυνση. Εμείς λέμε ότι η Τουρκία, ναι, έχει ρόλο στον ευρωπαϊκό χώρο. Εμείς λέμε ότι η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι, με μία όμως προϋπόθεση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι πρώτον να αναγνωρίσει ουσιαστικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Αν θέλετε έμμεσα να αναγνωρίσει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έδαφος πλέον ευρωπαϊκό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πολλά πρέπει να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και κλείνω όχι με το να καταθέτουμε απόψεις που ουσιαστικά είναι κατά της έννομης διεθνής τάξης και βεβαίως κατά του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτημένου. Ευχαριστώ. Merci. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Είναι πολύ σημαντική συζήτηση, αλλά μην επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο κυπριακό ζήτημα. Η κυρία Γιαννάκου που έχει δει στο λόγο και που είναι η σκιώδη συγγήτρια του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, ε, όταν σχολίασα την προσέγγιση του κυρίου Νταφ, για τον οποίο η εκτίμησή μου είναι ιδιαίτερη και η φιλία που μας συνδέει πολυετής, ε, βεβαίως δεν είχα υπόψη μου ότι ο κύριος Βανόρντεν θα έκανε όλα αυτά τα προσβλητικά σχόλια. Κύριε Πρόεδρε, με τη θεωρία του κυρίου Βανόρντεν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα βρει και με την Αλκάιντα και να συμφωνήσει και να είναι και από τις δύο πλευρές εξίσου υπεύθυνε σύμφωνα με αυτή τη θεωρία. Δεύτερον, ο κύριος Βανόρντεν λησμονεί ότι η χώρα του έχει μια τεράστια στρατιωτική βάση στην Κύπρο για την οποία κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης έθεσε θέμα πως αν δεν συζητηθεί πρώτα δεν μπει το πρωτόκολλο και δεν επαναληφθεί για τη Βρετανική βάση στην Κύπρο η Βρετανία αποχωρεί από τη συνέλευση και δεν συζητάει. Λοιπόν τα κρατικά συμφέροντα του καθενός τα ξέρουμε αλλά το να παρουσιάζεται εδώ μέσα όπως ελέγχθηκε πριν ο θήτης και το θύμα με τον ίδιο τρόπο είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δημιουργεί ανησυχία για το πώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι τη δημοκρατία και πώς διακρίνουν τη δημοκρατία από στενά συμφέροντα που πιθανόν να διακινούνται στη χώρα τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Euh, σας ευχαριστούμε ο κύριος και μετά ο κύριος Νταφ. Chairman, Πρόεδρε. Αυτή η ρήτρα αλληλεγγύης μας απασχολεί αυτή τη στιγμή και η γρήγορη ανταπόκριση. Αυτό είναι το θέμα του κυρίου Πάσκου. Αν είναι πραγματικότητα ή όχι αυτή η δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης σε περίπτωση επίθεσης κατά μίας χώρας μέλου καμίας και οποιασδήποτε. Εδώ χρειάζεται κάποια αποσαφήνιση στις παραγράφους 13 και 14. Γιατί καταρχάς φαίνεται να υπονοεί μόνο τρομοκρατικές επιθέσεις ή θεομηνίες. Η Ένωση τότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί. Το 14 όμως μας μιλάει και για ευελιξία ως προς τον ορισμό των τύπων επίθεσης για να διασφαλιστεί ότι καμία απειλή ούτε και οι κυβερνοεπιθέσεις δεν θα μένει αναπάντητη. Είχαμε δει περιπτώσεις επιθέσεων όχι μόνο κατά μεμονωμένων χωρών αλλά και της Ένωσης ολόκληρης και ηλεκτρονικός. Πριν από πολλά χρόνια θα θυμάστε την ηλεκτρονική επίθεση που έγινε κατά της Εσθονίας. Αλλά δεν δόθηκε καμία απάντηση από την Ένωση. Το ΝΑΤΟ ανησύχησε μόνο. Και η Ένωση έχασε εκεί την αξιοπιστία της γιατί δεν ενδιαφέρθηκε να μην επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις. Όταν βλέπω τις παραγράφους 15 και 16 διαπιστώνω μία βασική αντίφαση με τη 13 και 14 μεταξύ 13 και 14 από τη μία και 15 και 16 από την άλλη. Στο 15 και το 16 υπονοείται ότι ίσως να φταίει το θύμα. Γιατί πρέπει, χρειάζεται να αποδεικνύει εκείνο την ενοχή. Πρέπει λέει να αποδεικνύει μια χώρα που έχει τύχει επίθεσης ότι δεν έχει επαρκείς από μόνες της δυνατότητες ανταπόκρισης. Γιατί ζητάει αλληλεγγύη λοιπόν. Μήπως λέει δεν έχετε επενδύσει στην ασφάλειά σας επαρκώς. Ποιος θα κρίνει όμως αυτά τα πράγματα στο Συμβούλιο να κάνει την έρευνα να καταλήξει και τότε γιατί γρήγορη ανταπόκριση μιλάμε αν χρειάζονται τέτοιες έρευνες. Αυτά είναι γραφειοκρατία, διαδικασίες και οι ίδιες οι διαδικασίες μπορεί να αποτελέσουν καταστροφή. Πώς θα λυθεί αυτό. πρέπει να προσέξουμε αυτή την αντίφαση μεταξύ δύο και δύο παραγράφων. Μήπως πρόκειται εδώ για κάποια υποκρισία. που αντιφάσκει με την πραγματικότητα, που ε, η αντίφαση είναι μεταξύ λόγων και έργων. Υπάρχει και η έκφραση ότι η εφαρμογή της ρήτρα αλληλεγγύης πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα των διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων κλπ. Σωστό είναι, αλλά... Αλλά ακόμη και αν εννοούμε ότι η οι και οι θεομηνίες και οι καταστροφές οι ανθρωπογενείς καταστροφές τι σημαίνει. Μπορεί να είναι κρατικογενείς καταστροφές για κατά μίας γειτονικής χώρας. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορά μόνο κάποιους τρελούς αλλά και κάποιους τρελούς πολιτικούς καμιά φορά από γειτονική χώρα. Ε, και τώρα για την εφαρμογή που να είναι λέει αναπόσπαστο τμήμα της αντίδρασης κτλ. Καλή η πρόθεση μεν αλλά καταλήγει να μην οδηγεί η εφαρμογή στη δημιουργία ad hoc εργαλείων. Να μην οδηγεί. Αν δεν μπορούμε να δημιουργούμε ad hoc εργαλεία και μέτρα, τότε γιατί ανταπόκριση και απάντηση μιλάμε ιδιαίτερα δε ταχεία. ποια πραγματικότητα, μιλάμε για όνειρα. Είναι εδώ λεκτικά παιχνίδια και δεν επικρίνω εδώ τον κύριο Πάσκου, αλλά ίσως υπάρχει γενικά υπερβολική ευελιξία εδώ αν θέλουμε να συνδυάσουμε πραγματικότητες που υπάρχουν σε πολλές περιφέρειες με ευσεβείς πόθους. Μετά το 24 μας λέει ότι το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης ιδιαίτερα δύσκολων οικονομικών καταθάσεων. Όχι πρέπει, αλλά μπορεί. Μετά από μακρές συζητήσεις. Ε, τότε δεν μιλάμε πια για ταχεία ανταπόκριση. ιδιαίτερα αν υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην προμήθεια ορισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα ενεργειακών. Γιατί δεν λέμε τα πράγματα ρητά. Μπορεί να συμβεί να μπλοκαριστεί η προμήθεια ενεργειακών πόρων ως πολιτικό μέτρο. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική καταστροφή. Και μάλιστα μπορεί να γίνει αυτό και μόλις πριν από εκλογές. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Θα θέλαμε, αν και είμαστε μέλη της Ένωσης, να ακούσουμε ρητές και σαφείς θέσεις, όχι ασάφιες, με διατυπώσεις που να μπορούν να παρεμεινευθούν με ακριβώς όπως λένε με ευελιξία. Ίσως χρειάζεται λίγο λιγότερη ευελιξία εδώ στη διατύπωση και χωρίς υποκρισία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πιο σύντομες οι παρεμβάσεις σας και επικεντρωμένες σε συγκεκριμένο στόχο. Διαφορετικά δεν θα προλάβουμε κύριος Βανόρντεν επιθυμεί το λόγο μετά από όσα προηγούμενα υπόθηκαν. Σύντομα, σύντομα, ο κύριος Νταφ και ο κύριος Πασκού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να απαντήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις που με αφορούσαν για την Κύπρο. Ζητώ από τους συναδέλφους να ακούν αυτά που λέγω και όχι να φαντάζονται κάποια πράγματα. Πρώτον, μιλάμε για τις ε, βρετανικές βάσεις. Αυτό είναι κυριαρχικό βρετανικό έδαφος και δεν αφορά καθόλου τη διαφορά μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί. Τρίτον και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει την Προεδρία της Ένωσης τώρα έχει και ιδιαίτερη ευθύνη για να επιφέρει θετικές και επικοδομητικές αλλαγές αυτό θα έπρεπε να αποτελεί το μείζον επίτευγμα της Προεδρίας σας και τίποτα άλλο να μην κάνετε στην Προεδρία σας. Αυτό και μόνο θα αποτελούσε μια τεράστια επιτυχία. Αντίθετα όμως προτιμάτε να το παραμερίζετε και να λέτε δεν υπάρχει χρόνος για να συζητηθεί το θέμα στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Έχετε μεγάλη ευθύνη που νομίζω ότι δεν την αναλαμβάνετε σωστά. κλείνει η συζήτηση σχετικά με το κυπριακό θέμα και να επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική για την άμυνα κλπ. Να σας πω ότι ε, έχει αποδείξει ε, ότι διακατέχεται από ένα επικοδομητικό πνεύμα ακριβώ στην ε, διακοινοβουλευτική διάσκεψη πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο και ασχολείται, είχε το θάρρος να ασχοληθεί με δύσκολα θέματα όπως τις σχέσεις ε, με την Τουρκία και ότι τα θέματα αυτά δεν προσπάθησε να τα αποφύγει η Κυπριακή Προεδρία. Γι' αυτό θα, θα χαιρετήσω τις ε, προ Βουλίες ε, Ανδρίου. Δεν νομίζω ότι θα λύσει το Κυπριακό η έκθεση αυτή, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, μην το χειροτερέψουμε όλα στο Κυπριακό. με την ε, διατύπωση πιο συγκεκριμένης προσέγγισης από το Κοινοβούλιο στο θέμα της ε, αμοιβαία, της αλληλεγγύης. Ε, ε, η δική μου γνώμη, στην οποία εμένω, είναι ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα βοηθήσει την προσέγγιση προς μια επίλυση της ε, διέρεσης του νησιού και συμφωνώ με τον Τζέφρι Βαν Όρντεν στο βαθμό που δεν πιστεύω ότι η προσέγγιση συνοψίστηκε, που συνοψίστηκε από τον κύριο Σοφοκλέους ότι μπορούμε να περιμένουμε για μια λύση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Προς την κυρία Λέζινγκ θα έλεγα ότι ελπίζω η Γκουε να μην ε, διαβάζει από το Google για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχουν άλλες πηγές για να ενημερωθεί και μπορώ να συστήσω και άλλες πηγές εγώ ίδιος. Δεν είναι σόφρον να επιδιώκουμε να είμαστε υπερβολικά συγκεκριμένοι όταν μιλάμε για ορισμούς ειδών κρίσεων που θα ενεργοποιούσαν ενδεχομένως την ρήτρα αλληλεγγύης. Δεν αναζητούμε κάζους μπέλη εδώ. Εδώ ψάχνουμε πραγματιστικές, ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν ευέλικτες και ταχείες αποκρίσεις και ξεκάθαρα μέτρα και διοικήσεις και ελέγχους. Θα πρέπει να δημιουργηθούν όλα αυτά και θα πρέπει να υπάρχει έτσι δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια πληθώρα πολιτικών και στρατιωτικών απειλών. και καταστροφών. Ο Τζέφρι Ορντέν φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το έχει ξαναπεί. Να πω πάλι ότι το άρθρο 42.7 είναι άμεση αντανάκληση του άρθρου 5 της Συνθήκης των Βρυξελών της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πολύ σωστά συνοψίζεται. Ο κύριος Βανόρντεν, είμαι σίγουρος, δεν θα ήθελε να δει την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση να κολλήσει εργή και να παραμένει σε μία α στην οποία θεωρώ ότι είχε μείνει για πολύ μακροχρονικό διάστημα. Είναι σωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα μία πρόβλεψη για την αμοιβαία άμυνα ή αρρωγή, η συνδρομή. Αλλά η πρωταρχική θέση και το, ο, ο πρωταρχικός χώρος και το μέσον για την αμοιβαία άμυνα είναι όντως το ΝΑΤΟ. Θα έλεγα στην κυρία Γιαννάκου ότι με κατηγόρησε ότι παρουσίασα θέση βρετανική. Και ποια είναι η βρετανική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω. Και νομίζω ότι θα διέκρινε τουλάχιστον ένα ίχνος διαφωνίας μεταξύ του κυρίου Βανόρντεν και εμού, ώστε να υποπτευθεί ότι δεν υπάρχει βρετανική θέση ενιαία εδώ. Και προσβλέπω στο μέλλον να δω σαφέστερα πού ακριβώς επιλέγει να διαφωνήσει η κυρία Γιαννάκου με την προσέγγιση μου. Ναι, η Ευρωπαϊκή, ναι, η Επιτροπή, μήπως θα ήθελα να λάβει το λόγο, σύντομα όμως σας παρακαλώ, σχετικά με το θέμα αυτό της ελεγγύης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα σύντομα να πω εξ ονόματος της Κομισιόν ότι χαιρετίζουμε την έκθεση του κυρίου Πασκού είναι πολύ καλή η ισορροπία που έχει, αναγνωρίζει την παρούσα κατάσταση αλλά και τις βελτιώσεις που μπορεί και πρέπει να γίνουν. Θα εστιάσω τα σχόλιά μου στο άρθρο 222 και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό το άρθρο ε, θέλει να αποκριθεί και να βοηθήσει ε, στην αντιμετώπιση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι η ρήτρα αλληλεγγύης ε, που υπάρχει στη συνθήκη προσφέρει τρόπον την το νέο στοιχείο ώστε να επιβάλλουμε νομική υποχρέωση σε ένα κράτος, στα κράτη-μέλη να δράσουν από κοινού σε πνεύμα αλληλεγγύης μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Αυτή είναι νομική υποχρέωση, ήδη υπάρχει ε, ήδη είναι ενισχύει επί τη βάση της συνθήκης. Αυτό που ζητεί ε, περαιτέρω από την Κομισιόν και την ύπατο η εκπρόσωπο από κοινού η ε, συνθήκη είναι να υπάρξει πρόταση εφαρμογής των διατάξεων. Επί, επί της ουσίας της έκθεσης ευχαριστούμε τον κύριο Πάσκου και την Επιτροπή εδώ διότι προσφέρουν και παρουσιάζουν πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις που, με τις οποίες συμφωνούμε, όπως ότι πολλά μέσα υπάρχουν ήδη στη διάθεσή μας σήμερα και μπορούν να συμβάλλουν για να αντιμετωπιστούν τα μετέπειτα τέτοιων καταστροφών. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει συνοχή, να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και επίσης εκτιμούμε ε, την υποστήριξη μέσα στην έκθεση για την πρόταση, για παράδειγμα, ε, για καινοτόμα στοιχεία στην πολιτική προστασία. Ε, Αυτό είναι ένας τομέας βέβαια που αποτελεί έναν από τους κέριους πυλώνες για την εφαρμογή της ρήτας αλληλεγγύης. Επίσης σημειώνουμε την πρόθεση ε, να συνεχιστούν εργασίες σε άλλους τομείς όπως εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, ενημέρωση με πληροφορίες, ε, παρακολούθηση εκθέσεων ε, κινδύνων επικινδυνότητας, ε, ε αντίκτυπου επικινδυνότητας, ανάλυση επικινδυνότητας. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την επικουρικότητα, την ελευθερία που έχουν επιλέξει και διαδηλώσει στη συνθήκη τα κράτη-μέλη. Σταματώ εδώ για να πω ότι η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να επεξεργαστεί μια κοινή πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου πάνω στο θέμα αυτό και ελπίζομαι να την παρουσιάσουμε πριν από το τέλος του χρόνου. Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμβολή στην προβληματική μας σε αυτά τα θέματα και προφανώς θα κρατούμε το Κοινοβούλιο πλήρως ενημερωμένο για την πορεία των ε, εξελίξεων. Σας ευχαριστούμε υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Για να δούμε κάποιος μήπως θα επιθυμούσε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου. Επιβεβαιώνω δηλαδή ότι δεχόμαστε την έκθεση του κυρίου Πάσκου που τη βρίσκουμε επίκαιρη και χρήσιμη. και συμφωνώ με τους άλλους συμβοναδέλφους της Κομισιόν ή της Επιτροπής ότι πρέπει το σύστημα που θέλουμε να δημιουργήσουμε να έχει ταχεία ανταπόκριση σε καταστροφές με πλήρη σεβασμό της ρήτρα αλληλεγγύης. Να είναι συνεπές, αποτελεσματικό, να αποφεύγει τις επικαλύψεις και είμαστε βέβαιοι ότι οι υπάρχουσες δομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκεί να συντονιστούν καλύτερα και να υπάρξει έτσι ένα ισορροπημένο σύστημα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις μεγάλων διαστάσεων καταστροφών. Φυσικά δεν αγνοούμε την πολιτική διάσταση όλων αυτών, το ποιος θα αποφασίζει και πώς θα ταυτίσουμε πότε αρχίζει να ισχύει η ρήτρα αλληλεγγύης. Αυτό φυσικά δεν υποκαθιστά καμία άλλη αντίδραση της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 34 και η έκθεση του κυρίου Πάσκου αυτό λέει. Τέλος. γνωρίζουμε ότι πρέπει να ταυτίσουμε καλύτερα ποιες ακριβώς πρέπει να είναι οι δομές που θα συντονιστούν. Ευχαριστώ. Καταληκτικά τώρα ο κύριος Πασκού, εισηγητής, και να πενθυμίσουμε κάτι ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες έχει οριστεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Κανονικά ήταν στις 20, πήγε στις 21 τώρα και 9 Οκτωβρίου για μια νέα συζήτηση που θα συμπεριλαμβάνει και τις τροπολογίες. Ευχαριστώ όλους. γιατί εξετάσατε πολύ σοβαρά την έκθεση. Αναφέρατε και σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν ή να έχουμε περισσότερη ανάλυση τους. Οι παράπλευρες πολιτικές συζητήσεις που έγιναν εδώ δείχνουν επίσης ότι πρόκειται για έκθεση όπου πρέπει να προσέξουμε πολύ. Το ξέρουμε. Δεν θέλουμε να θίξουμε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να μπορέσουμε με την απέξω, για να το πω έτσι, άποψή μας στην επίλυση προβλημάτων. Η Ένωση είναι νομοθετικό σώμα με βάση τη ρωμαϊκή παράδοση του δικαίου κτλ. εμείς τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση τη συμπεριλάβουμε στη συνθήκη. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί μια χώρα να ζητήσει την ενεργοποίηση της ρήτρα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ, γιατί να συζητιούνται πρώτα τα πράγματα στην Ένωση και μετά να βλέπουμε αν χρειάζεται να προσφύγουμε στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, από την εμπειρία μου έμαθα ότι όσο πιο ακριβείς είμαστε στη διατύπωση, τόσο λιγότερα αποτελέσματα έχουμε στην πράξη. Η ευελιξία είναι κάτι πολύτιμο γιατί τελικά, τελικά όλα μπορούν να τύχουν ερμηνείας και παρερμηνείας. Το ΝΑΤΟ ας πούμε που στο άρθρο 5 γίνεται λόγος για αυτόματη ανταπόκριση κλπ. Ναι μεν αλλά πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για θέμα του άρθρου 5 για την Τουρκία και τα Άγουαξ με το Ιράν χρειάστηκαν 11 μέρες. Εν τω μεταξύ όμως υπάρχει η απειλή. Κύριε Λαρμπέντζη λοιπόν, Λαντσμπέργκης μάλλον, καταλαβαίνω τι εννοείται αλλά είναι μάταιο να λέμε στο Συμβούλιο πρέπει αντί για μπορεί θα ε, μπορούσε γιατί το Συμβούλιο ούτως ή άλλως θα κάνει ό,τι θέλει. Ενώ στο ΝΑΤΟ τα σημαντικότερα πρόσωπα είναι οι εκπρόσωποι των χωρών επίσης, οι οποίες χώρες όπως και στο Συμβούλιο πάντα βρίσκουν τρόπους να προστατέψουν το εθνικό του συμφέρον. Η ελαστικότητα λοιπόν λειτουργεί και υπέρ ημών γιατί μας επιτρέπει να φέρουμε στην τράπεζα των συζητήσεων θέματα που αλλιώς αν είμαστε πολύ αυστηρά διατυπωμένοι θα μας πούν ότι δεν καλύπτονται ακριβώς αυτά τα θέματα από τη διατύπωση λοιπά. Είπατε επίσης ότι δεν θέλουμε να δημιουργούνται ad hoc εργαλεία. Ναι. Ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τη δημιουργία νέων οργανισμών. Θα είναι φωνή όντως εν τη ερήμα. Και δεύτερον, υπάρχουν αρκετά εργαλεία και μέσα και πρέπει καταρχήν να φροντίσουμε να λειτουργούν με πιο συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο. Και μετά να δούμε τι μπορεί να παραλείπεται και μπορεί να χρειαστεί να δημιουργείται. Αυτά είχα να σας πω. Χαίρομαι που παρατάθηκε η διορία κατάθεσης τροπολογιών. Στις 20 θα συνεννοηθούμε και με την Κομισιόν. Είναι ρευτά τα πράγματα αλλά η πόρτα είναι ανοιχτή. Αν έχετε προτάσεις μέσω τροπολογιών ή αλέως, με τα χαράς να τις ακούσουμε. Κύριε Σιγητά. Αυτός ο συνδυασμός και των ακαδημαϊκών εμπειριών σας και των πρακτικών ε, επιχειρημάτων σας τα κάνουν όλα να είναι πραγματικά συμπαθητικά και είναι κάτι το ρεαλιστικό και στον τομέα αυτό όπου η εθνική κυριαρχία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη, χρειάζεται ιδιαίτερος ρεαλισμός για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ο δογματισμός δεν μας κάνει να προχωράμε και τόσο πολύ σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε επιλέξει. Σας ευχαριστούμε για τη σημαντική αυτή συζήτηση. Θα συνεχιστεί μετά στις 9 Οκτωβρίου μετά από την καταστροπολογιών. Ευχαριστούμε, Άντριο, για την βοήθειά σας και από τη συνεργασία μας αυτή. Είμαστε σίγουροι θα έχουμε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο, καλό, θετικό κείμενο σαν έκθεση και ο Συμβούλιο, Πρόεδρος Συμβουλίου ε, έχει σαν πρόθεση τα θέματα άμυνας να τα συμπεριλάβει από το Δεκέμβριο ήδη στην ημιστή διάταξη και την άνοιξη στη συνέχεια και πάνω σε αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα ε, να μπορέσει να βοηθήσει με τη σοφία το Κοινοβούλιο μέχρι τότε και με την ψήφιση τον Νοέμβριο και τώρα για την αλληλεγγύη αυτή, τον Οκτώβριο για το θέμα ένα διαλυματάκι δύο λεπτά σας παρακαλώ και θα επανέλθουμε με το PSDC με την ετήσια αυτή έκθεση. Ευχαριστώ. Bien, chers collègues, si nous pouvons reprendre. Merci de regagner. Παρακαλώ στις θέσεις σας και πάλι. Το πρώτο μέρος για την Uh, εφαρμογή της κυρίας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ε, και όπως έχει οριστεί από το Προεδρείο ε, εγώ θα έχω αναλάβει το θέμα αυτό. Έχουμε αρκετά σημεία. Να σα υπενθυμίσω μερικά πράγματα. Χρειάζεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια, όπου θα είναι και ε, η υπεύθυνη ύπατος αρμοστής ε, της 26 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον ένα μήνα, αλλά θα πρέπει όμως να εργαστούμε αρκετά γοργά δεν έχει και μεγάλες εκπλήξεις σε σχέση με προηγούμενα που έχει οθετήσει το Κοινοβούλιο. λοιπόν, οι συζητήσεις κανονικά δεν θα πρέπει να διαρκέσουν και πολύ γιατί γνωρίζουμε αρκετά καλά τις θέσεις των ομάδων, γνωρίζουμε ποια σημεία δημιουργούν ε, περισσότερα θέματα, προβλήματα, εντάξει θα δούμε και θα πρέπει να εργαστούμε αρκετά γοργά και ναι, σύντομα ώστε στις 26 Οκτωβρίου να είμαστε θέση να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση και ίσως η έκθεση θα ήθελα να πάει παραπάνω από μερικές διαπιστώσεις όπως κάνουμε συνήθως. Σίγουρα έχουμε 15 αποστολές ε, που ισχύουν πάντα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής και ο στόχος ε, της έκθεσης είναι να εξετάσουμε τις στρατιωτικές και πολιτικές αυτές αποστολές, ποιες είναι αποτελεσματικέ, ποιες όχι, σε όσες είναι λιγότερο αποτελεσματικέ, να κάνουμε συστάσεις, αυτές είναι ο πρώτος μας. Αλλά πέρα λοιπόν από διαπιστώσεις επιτόπου, σύμφωνα με όσα έκανε και ο συνάδελφος της Μπροκ ε, για την ΠΕΣΚ, εδώ θα πρέπει να δούμε σε ποια πλαίσια αυτή η πολιτική ασφαλείας και άμυνας ασκείται και η συνήθειά μας είναι να εργαζόμαστε βασιζόμενοι στην στρατηγική για την ασφάλεια του 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναθεώρηση το 2008 αλλάζουν ε, οι συνθήκες και πολλά αλλάζουν από πλευρά στρατηγικής πολιτικής ε, και θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία και υποχρεώσεις που προκαλούν λαγές σε αυτή την πολιτική. Σίγουρα είναι οι ανοιχτές κρίσεις πάντα, είτε οι τεταμένες σχέσεις και στη Μέση Ανατολή και το Μεσοβορανότο και είναι σημαντικές κρίσεις γιατί οι εξελίξεις ε, ίσως ε, είναι θετικές, αλλά ίσως ε, δημιουργούν και έλλειψη σταθερότητας και μας κάνουν ανησυχούμε ε, για την κατάσταση στο νότο μας, όπως στη Λιβύη, ε, και στη Λιβύη και στη Συρία τώρα, αλλά σίγουρα και όλη αυτή η μεταβατική περίοδος σε αραβικές χώρες, την Ισία, Αίγυπτο και αλλού, και οι σχετικές εξελίξεις δημιουργούν προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά θέματα ασφάλειας επειδή όλο και περισσότερο εξαπλώνται και τα πυρηνικά όπλα, να σκεφτούμε την ε, Ιρανική περίπτωση, εδώ είμαστε σε κρίσιμη φάση, γιατί είναι μεγάλες οι απειλές ε, και έχουμε διάφορες δυνατότητες είτε διπλωματικής φύσεως είτε στρατιωτικής φύσεως ε, που θα επηρεάσουν έντονα την κατάσταση και πέρα από αυτό και την ασφαλεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ παίζει ρόλο όμως και ένας παράγοντας που δεν έχουμε λάβει τόσο υπόψη μας ίσως μέχρι τώρα, ο επαναπροσανατολισμός ο στρατηγικός των Αμερικανών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, το είδαμε άλλωστε στην ετήσια έκθεση, ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα το ανέφερε, θεωρούν ότι αυτό που έχει προτεραιότητα στην άμυνα εξασφάλεια για τα συμφέροντά τους είναι στην Ασία και στον Ειρηνικό. Είναι νέα σχετικά στοιχεία. Έχουμε συνηθίσει εμείς οι Ευρωπαίοι έτσι, με την άνεσή μας να απασχολούμε εμείς τους Αμερικανούς είτε στην στα στρατιωτικά μας τμήματα, στρατεύματα, είτε και σε σχέσεις μας ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια δεν είναι ότι αμφισβητούν τώρα πια για τις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ αλλά είναι νέα διαθωτικά στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, σε σχέση με όσα θέλουμε να κάνουμε για την ε, ε, κοινή στρατηγική πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Αυτά θα ήθελα να προσθέσω κάτι και την οικονομική κρίση σε κονδύλια, στον προπολογισμό παντού, σε όλα τα κράτη χωρί καμία εξαίρεση Ευρωπαϊκής Ένωση, σε όλα τα κράτη μειώνουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Ευτυχώ έντονη αυτή η τάση, διαφορετικό το θέμα, δεν είναι μόνο συγκυριακό ε, και θα πρέπει να το συνηθίσουμε, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και όλη η αρχιτεκτονική της κοινής πολιτικής φοράς και άμυνας ε, όπως επηρεάζονται από θέματα προπολογισμού. Αυτές οι νέες ποιώσεις που επηρεάζουν αυτή την κοινή πολιτική και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Βέβαια θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι εδώ δεν είναι μόνο να δούμε ποιες είναι οι μη ρεαλιστικές μας φιλοδοξίες για την αυτή κοινή πολιτική ασφαλής και άμυνας και να θέλουμε έτσι ιδεαλιστικά και μόνο ένα ποιοτικό άλμα, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι από τις συνθήκες της Αβώνας και μετά έχουμε μέσα εργαλεία και πριν από τις ειδήσεις της Αβώνας είχαμε μια κάποια οργάνωση από το 1999 ορισμένα όργανα που, εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι για δύο κυρίως λόγους Δηλαδή, επειδή ε, έχουν μια κάποια διστακτική στάση τα κράτη και μια κάποια απάθεια, αδράνεια των ε, οργανώσεων ε, υπό την κυρία Άστον ε, Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούνται όπως πρέπει, όσο πρέπει κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και από τις κρίσεις εδώ κοντά μας. Το είδαμε, το είδαμε με τη Λιβύη και το βλέπουμε και σήμερα με τη Συρία και στην περιοχή του Σαχέλ ε, βλέπουμε τι γίνεται, ότι υπάρχουν ε, δυσκολίες να την ασφάλεια κλπ. Αυτή η δυνατότητα για ειρηνευτικές ενέργειες έχει υποχρησιμοποιηθεί. Ε, δεν θα πρέπει να τεινωθούμε την κοινή αυτή πολιτική άμεση να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει, δεν είναι εργαλείο κοινή άμυνα, αλλά θα πρέπει να μπορεί να παίξει το ρόλο που έχει και που έχει επισημοποιηθεί από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτά υπενθυμίζει και η έκθεση αυτή και θέλουμε έτσι να συνειδητοποιήσουν τα κρατημέλη και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα εργαλεία ήδη μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Αυτό ισχύει και από πλευράς βιομηχανίας. Βλέπουμε τις εξελίξεις λόγω της δυσκολίας της οικονομικής. Θα πρέπει να δούμε το ρόλο που θα παίξουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον όλο ορισμό της ε, βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας και να δούμε το ρόλο που θα επιθυμούμε να παίξουμε. Είναι ανοιχτοί λοιπόν δρόμοι που προτείνονται όπως και κάθε χρόνο δε. Έχουμε τομεί όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα επιμένει μια λευκή βίβλο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη βιομηχανική τεχνολογική Ευρωπαϊκή Βάση και Ίσως θα πρέπει να δούμε μια κοινοτική προτίμηση γιατί έχουμε να κάνουμε με τη βιομηχανία άμυνας που είναι μια δύναμη εκεί ευρωπαϊκή δεν θα παραμείνει αν δεν ασχοληθούμε και υπάρχουν και προκλήσεις τεχνολογικές και απασχόληση και επίσης έχουμε και τώρα από κοινωνική πλευράς θέμα θα πρέπει να δούμε αν η Ευρώπη θα επιθυμεί να είναι ανταγωνιστική ήπειρος στα θέματα αυτά, στο αυτούς επίσης η διαστημική πολιτική, σημαντικά θέματα και επίσης να δούμε ένα κάποιο προγραμματισμό. Ήδη συζητήσαμε γι' αυτό με την έκθεση Πασκού, αυτό το γενικό επιτελείο το επιχειρησιακό, το οποίο συζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια, ξέρουμε ποιοι είναι αντίθετοι, πώς είναι αντίθετοι, πάντως ε, δεν θα πρέπει να ε, αποσυρθούμε από αρκετά από αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτή είναι η συζήτηση και επιμένω γιατί ε, τα είδαμε, τα συζητήσαμε αυτά πριν από δύο χρόνια και θα ήθελα να επιμείνω στο εξή. Ένα από αυτά που συνέχεια μας απασχολούν είναι η στρατηγική αυτονομία η φιλοδοξία για κάτι τέτοιο εδώ. Δεν φτάνει να πούμε ότι θα πρέπει να κάνει τα πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της και τα πάντα και εις βάρος των, ε, των, των, ε, των συμμαχιών, ε, δηλαδή εις βάρος του ΝΑΤΟ ας πούμε, αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να μπορεί να πει όχι σε αποφάσεις που την αφορούν, αλλά δεν υπήρξαν οι σωστές συζητήσεις και είδαμε και στο παρελθόν από ορισμένους από τους συμμάχους μας να παίρνουν ε, ε, μονόπλευρα αποφάσεις και να δούμε πώς η Ευρώπη θα μπορούσε και από μόνη της να παρεμβαίνει εκεί που διακυβεύονται συμφέροντά της αλλά και εκεί που οι συμμαχοί της εκτός Ευρώπης για διάφορους λόγους δεν θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν. Θα πρέπει να φυλάξουμε τα συμφέροντά μας και εκεί ακριβώς που θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Αυτό εννοούμε σαν στρατηγική αυτονομία και πέρα από μια ισχυρή κατάσταση που νομίζω ότι στα υπόλοιπα συμφωνούμε. Σίγουρα θα έχουμε μια ευρεία συζήτηση πάνω σε αυτό και εντάξει όχι από κακόπιστα αλλά μετά από όλα αυτά που βλέπουμε στρατιωτικοποιείται η... νομίζουν ορισμένοι η πολιτική αυτή όχι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο απλά και μόνο θέλουμε να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει στο σύνολό του πλήρως το εργαλείο αυτό και ένα μικρό μέρος των εργαλείων που διαθέτουμε είναι ε, από πλευρά στρατιωτική πτυχής ακριβώς και είναι και το τελευταίο στο οποίο πρέπει να καταφύγουμε. Δεν είναι απόλυτη προτεραιότητα, αλλά την στιγμή που θα χρειαστούμε αυτά τα εργαλεία, αν δεν τα έχουμε φροντίσει, αν δεν τα έχουμε λάβει όπως πρέπει υπόψη μα ετοιμάσει, προετοιμάσει προσωπικό, ε, εργαλεία, θεσμική δυνατότητα λήψη αποφάσεων, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και μην ξεχνάμε αυτό που έγινε σχετικά με την λιβική κρίση. Δεν μπορούσαμε να δούμε όπω πρέπει, γιατί είχαμε ξεχάσει πώς να τα χρησιμοποιούμε. Δεν μιλάμε για παρέμβαση, μιλάμε για σχεδιασμό δεν είναι ότι γλιστράμε προς ε, το στρατιωτική πτυχή, αλλά εδώ υπάρχουν όμως τα στρατιωτικά εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησαν εδώ και 10 χρόνια και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό το comprehensive approach, κατανοητική προσέγγιση δηλαδή, με προσέγγιση με κατανόηση και να δούμε την ε, προσθέμενη αξία της Ευρώπης αυτό και αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει και με τα στρατιωτικά εργαλεία, διαφορετικά δεν είναι συνολική σφαιρική προσέγγιση. Δεν θα είμαστε πια ανταγωνιστικοί από τη στιγμή που δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πτυχές αυτών των εργαλείων. Αυτή είναι η φιλοσοφία που διακατέχει την έκθεση και περιμένω τώρα να προσθέσετε στοιχεία, να βοηθήσετε, ελπίζω και είμαι σίγουρος μάλλον ότι το πνεύμα θα είναι επικοδομητικό στην όλη συζήτηση ώστε η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα ασχοληθεί το Συμβούλιο από το Δεκέμβριο με θέματα άμυνας και μετά ξανά το Άνοιξη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ θα πρέπει με τη σχετική αυτή ευκαιρία να δείξει ότι δεν καθυστερεί στην αντίδρασή του, ότι διαθέτει προτάσεις επικοδομητικές σε αυτά τα λεπτά ευαίσθητα θέματα και νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπερισχύσει ο ρεαλισμός γιατί οι διάφοροι αρνητικοί δογματισμοί ή ιδιαίτερα μεγάλος μεγάλη ευαισθησία με ιδεαλισμό. Αυτό δεν βοηθάει αυτά. Ο κ. Γιάννης ε, έχει το λόγο. Σκιώδης συγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ γιατί είστε εισηγητής ε, στην σημαντική αυτή έκθεση όπως επίσης και γραπτά και προφορικά για το σε ποια σημεία επικεντρώνει την προσοχή σας ε, που έχει να κάνει με τα βασικά σημεία που έχουν επηρεάσει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, και ταυτόχρονα με συστάσεις προς την υπατορμοστή μας την κυρία Άστον για να βελτιωθούν τα πράγματα σε σχέση και με τις προκλήσεις. Ε, είχαμε παρόμοιες εκθέσεις, δεν ξέρω αν χρειάζεται τώρα όμως να τα πούμε. Είχαμε πει ότι οι μεγαλύτερες ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο ότι απέναντι σε μια κάποια κριτική που ασκείται θα ήθελα να πω κάτι που σε εκείνους μέσα στο κοινοβούλιο κρατούν μια εθνικής, ιδιαίτερα εθνικής φύσεως για την κυρίαρχη θέση, εθνική κυριαρχία και οποιαδήποτε πρόοδος σε κοινέ πολιτικές, κυρίως σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, τους καθιστά νευρικούς και προκαλεί την ευρικότητά τους ακριβώς και με προβλήματα στη χώρα τους, αν είναι μεγάλη χώρα τους. Αλλά επαναλάβαμε πολλές φορές ε, όλα αυτά δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις και στον κόσμο και στην Ευρώπη. Δεν μιλάμε για μια συγκεκριμένη χώρα, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε πάντα όλα αυτά στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αυτά τα πράγματα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε πάντα σε βάθος, σε λεπτομέρειες, ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είναι ένωση, όπω το όνομά της, το έτσι, έτσι θα πρέπει να συνεχίσει. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα προκύψει ακριβώς όταν μιλάμε για παρόμοια θέματα. Πρέπει να βρούμε αυτό τον ε, ειρηνικό μηδενισμό και όταν μιλάμε για εργαλεία άμυνας και ασφάλειας ε, θεωρούν ότι σώνει και καλά θα πρέπει να είναι μια στρατικοποιημένη Ευρώπη. Όχι, όχι επαναλαμβάνω. Απλά και μόνο χρειάζεται να μπορούμε να προσφύγουμε στα εργαλεία που διαθέτουμε όταν χρειάζεται ε, δυστυχώς καμιά φορά για να εγγυηθούμε την ασφάλεια, την άμυνα, την ειρήνη των συμπολιτών μας και έστω και αν αυτό απαιτεί ορισμένα πράγματα όπως στρατιωτικοποίηση και μια επιθετική πολιτική και η πολιτική πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται, βασιζόταν πάντα σε αμυντική πολιτική προστασία και όχι επίθεση Ακόμα και τώρα τους τελευταίους μήνες που έγινε της μόδας παρόμοιο επιχείρημα με... για τη Λιβύη και στη συνέχεια κάτι παρόμοιο που θα έπρεπε να γίνει στη Συρία. Εμείς ε, που είμαστε πέστης παίξ, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες ε, που είχε και θα έχει και στο μέλλον οποιαδήποτε παρόμοια ευρωπαϊκή παρέμβαση είτε από πολλές χώρες, ε, σε χώρα όπως τη Συρία, σε μια τόσο δύσκολη περιοχή και σε τόσο δύσκολη κατάσταση όπως την αντιμετωπίζουν εκεί. Θα πρέπει να δούμε αυτόν τον τομέα, αλλά υποστηρίζουμε τον εισηγητή ότι η πρώτη ευρωπαϊκή πολιτική με το 2003 με το Χαβιέ Σολάνα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει αρνητικά ή θετικά όσον αφορά πολλές πτυχές. Δεν υπήρχε τότε τόσο ιδιαίτερη οικονομική κρίση όπως τώρα σήμερα για αρκετές χώρες μας ούτε ο ριζοσπαστικός ε, Ισλαμισμός ε, Εξαπλώνονταν τόσο ε, σαλαφισμός από τη περιοχή της Αχέλ μέχρι την υπόλοιπη Αφρική και που επηρεάζει τα πράγματα με επιθέσεις εναντίον πρεσβειών ευρωπαϊκών και αμερικανικών. Βέβαια, υποστηρίζουμε την οικονομική πολιτική όπως μας το είπε ο Πρόεδρος μας, αλλά θα θέλαμε ταυτόχρονα να μπορέσαμε να ενισχύσουμε την πτυχή αυτή της πολύπλευρης αντιμετώπισης ε, κάτι με το οποίο ασχοληθεί τότε και θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε σε βάθος και με λεπτομέρειες ε, και θα δούμε μια δεχόμενη τροπολογία για την ευθύνη, για την προστασία και μέσω των εθνών καμιά φορά έχουν αντιδράσει σε αυτό και να δούμε για την σωστή εφαρμογή που είναι κάτι το προχωρημένο, προοδευτικό, όχι μόνο σε γενοκτονίες, σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και γενικά σε ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης την ανθρώπινη ασφάλεια. Θα ήθελα εκεί να δούμε περισσότερο και καλύτερα την αναφορά στους μισθοφόρους ε, ιδιωτικά σώματα ασφαλείας ε, στις, ε, στις νέες πολέμους γιατί από ό,τι βλέπω πολλές φορές όταν μιλάμε για ασφάλεια και άμυνα όπως και τώρα που έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στην ασφάλεια των κοντινών περιπτώσεων, ενώ θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε την ασφάλεια και σε μακρινές γεωγραφικά περιοχές, επειδή βλέπουμε μια στρατικοποίηση πολλών χωρών στην Ασία, ας πούμε, και κυρίως της Κίνας και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει τώρα που βλέπουμε τις σχέσεις Ευρώπης και Ασίας σε θέματα πολιτικής, κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα, αλλά προς το παρόν διακόπτω εδώ και θα ε, προσπαθήσουμε βέβαια όλοι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση που μας είπε ο πρόεδρος μας. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε την έκθεση ισορροπημένη, ρεαλιστική, πραγματιστική. Χρειαζόμαστε τέτοιο ρεαλισμό αφού ζούμε μια κρίση που εμποδίζει την εφαρμογή πολλών καινοτικών προγραμμάτων και να δούμε τα πράγματα σφαιρικά πρέπει να την στηρίξουμε όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις και γι' αυτό είμαστε υπέρ. Επειδή είμαστε φιλοευρωπαίοι υποστηρίζουμε όλα όσα είπε ο εισηγητής και πιστεύουμε ότι πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η σωστή εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι πιο εύκολο να διορθώσουμε και να συντονίσουμε τα υπάρχοντα όργανα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε για την πολιτική κοινή άμυνα. Επίσης για τις στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις πρέπει να θίξουμε το θέμα της ασφάλειας στο Μαλί όπου έχουμε αποστολή αλλά και στη Συρία. Δεν ξέρω αν είναι η καταλληλότερη στιγμή να τα πούμε εδώ, αλλά ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο και εκεί. Για τις δυνατότητες που έχουμε, στην έκθεσή μας όπως και στη δική σας, μιλάμε γι' αυτό, γενικά όμως έχουμε κοινή, κοινό όραμα και άποψη. Μόνο ένα έχω να προσθέσω, την αναγκαιότητα αναθεώρησης της στρατηγικής μας. Γιατί αλλάζουν σήμερα τα πράγματα ως προς την ασφάλεια, η κατάσταση είναι πολύ ρευστή και χρειαζόμαστε μία πιο ευέλικτη στρατηγική ασφαλεία στην Ευρώπη, ενημερωμένη με συμμετοχή όλων των χωρών. Τέλος, το θέμα των τροπολογιών. Ποια είναι η προθεσμία 21 Σεπτεμβρίου λίγη. Μάλιστα. Θα καταθέσουμε μερικές τροπολογίες κι εμείς. Ευχαριστούμε η κυρία Κρόνμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μ' αρέσει η δομή της έκθεσης. Είναι ένα σημείο φετηρίας με ρεαλισμό, χωρίς να θέλει τη στρατιωτικοποίηση της Ένωσης, αλλά αξιοποιώντα τα υφιστάμενα μέσα. Καλό λοιπόν το σημείο φετηρίας. Τώρα για τη Λευκή Βίβλο. Από το 2003 και το 2008 άλλαξαν τα πράγματα. Και αν επρόκειτο κανείς να ορίσει τις πιο σοβαρές απειλές ε, κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας ε, είναι η διάδοση των πυρηνικών στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα αν αυτό γίνει μετά από στρατιωτικό πλήγμα. Χρειάζονται ρεαλιστικά σενάρια λοιπόν στη Λευκή Βίβλο και να ξέρουμε ποιες ικανότητες θα χρησιμοποιηθούν σε ποιες περιστάσεις. Αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη υποστήριξη των λαών μας ε, για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, θα είναι σημαντικό βέβαια ο κόσμος να μπορεί να συζητεί τις σχετικά, τα σχετικά σενάρια απειλών που υπάρχουν και η συζήτηση πρέπει να γίνει με τρόπο κατανοητό. Τώρα για το pooling and sharing πρέπει να αρχίσουμε με τα 11 έργα, 11 από 300 ήταν αυτά που ξεκίνησαν και εδώ χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό πλαίσιο ώστε να είναι σαφές στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν σε ό,τι αφορά τη συνένωση των πόρων και το μοίρασμα των πόρων, για να υπάρχει εκεί πρόοδος. Τώρα, για τους βασικούς στόχους τους πολιτικούς, θα πρέπει να προωθηθούν. Χρειάζονται επίσης δεξιότητες διαμεσολάβησης. Είναι σημαντικό αυτό για να υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι δεξιότητες χρειάζονται και στην πρόληψη και στην οξία κρίση. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε το ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπαιδεύουν τον κόσμο, τουλάχιστον στη χώρα μου. Είχαμε συζητήσεις για την αστυνομία και την εκπαίδευση των αστυνομικών για τις πολιτικές αποστολές και ίσως αυτό θα πρέπει να γίνει ευρύτερα. Τέλος, για το σχεδιασμό. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη μόνιμης έδρας, μόνιμης διοίκησης για τον ε, στρατιωτικό σχεδιασμό να μην είναι σε βάση ad hoc. Ένα σημείο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι το πολιτικό σκέλος πρέπει να διαχωριστεί. Λειτουργεί καλά σήμερα. Αν έχουμε δύο μόνιμες διοικήσεις, ελπίζω ότι θα ενισχυθεί και η συνεργασία μεταξύ τους. Τέλος, για το θέμα των ε, μάχημων ομάδων, battle groups, ήμουν πολύ υπέρ και ήλπιζα πολλά και στη φιλανδική ομάδα για την άμυνα, αλλά αφού υπάρχουν δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται κιόλα. Δεν είναι επιχείρημα υπέρ τη χρήση. Καλό είναι να νιώθουμε ότι, έχουμε, ότι έχουμε τι μάχημε ομάδε, αλλά ε, μόνο αν χρειάζεται θα χρησιμοποιούνται. Δεν θα πάμε σόνι και καλά να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, αν ε, χρειάζεται, τότε ναι. Επίσης, ε, οι χώρες, ε, πρέπει να πούμε, πρέπει να σέβονται τις δεσμεύσεις τους. Πολλές σκανδιναβικές χώρες ε, τις σέβονται. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια περίπτωση που μπορούμε να το ξαναπούμε αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Λόζινγκ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή και ιδιαίτερα ευχαριστώ για τις επεξηγηματικές ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Μία προκαταρκτική παρατήρηση από μένα. Η θέση μου δεν πρέπει να ε, θεωρηθεί εθνικιστική. Είναι ε, περίεργο να μιλάμε για μηδενισμό. Ε, ε εμείς δεν το κάνουμε. Κύριε Ντανζάν είπατε ότι δεν ε, κατανοείτε την έκθεση αυτή ως ε, μια ενίσχυση του στρατιωτικού προσανατολισμού. Στη βασική έκθεση το βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα γιατί πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή είναι στο άνω όριο του φάσματος στρατιωτικού προσανατολισμού. Επίσης, θα υποβάλλουμε και εδώ μια έκθεση μειοψηφία και θέλω να διευκρινίσω αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα. Βρίσκω αξιοσημείωτο πόσο ενισχυμένος είναι ο προσανατολισμός στην Αφρική. Δεν το αξιολογώ αυτή τη στιγμή, απλώς το επισημαίνω. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν περιγραφεί κάποια ε, αυτόνομα, αυτο, κάποιες αυτόνομες ε, πτυχές ε, της ε, πολιτικής της Ένωσης. Άλλωστε είπατε και εσείς εισαγωγικά ότι αυτό είναι πολύ έντονο, και, ότι αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση με οικονομικά συμφέροντα. Να το εξηγήσετε καλύτερα. Αναφερθήκατε πολύ και στην κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη στα ίδια πλαίσια. Με ενδιαφέρει να μου πείτε πόσο συνδέονται αυτά με ένα στρατιωτικό προσανατολισμό. Θυμίζω δε ότι στην ε, Γερμανία ο πρόεδρος Κέλερ εξαναγκάστηκε σε παρέτηση ε, όταν ε, μίλησε για την υπεράσπιση της γερμανικής βιομηχανίας. Θέλω να παρατηρήσω άλλη μια φορά Ε, την σημασία της θέσης αυτής. Επίσης, είναι ενδιαφέρον, κύριε Ντανζάν, ότι στην έκθεσή σας, που είναι σχέδιο έκθεσης, ε, μιλάτε όμως ε, στηριζόμενος στην πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Μάλλον δεν λέτε την πλειοψηφία, λέτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί πριν από κάθε συζήτηση. Ακόμα και αν ληφθεί απόφαση κατά πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν παρόλα αυτά διαφορετικές απόψεις, αντιπολιτευόμενες. Οπότε αυτό το ερμηνεύω σαν κάτι καινοφανές, μια δημοκρατική διατύπωση που μέχρι τώρα δεν την έχω διαβάσει σε καμία έκθεση που να προδικάζεται τόσα πολλά πράγματα. Επίσης δεν συμφωνώ με τη λογική συναδέλφων και τη δική σας λογική ότι ένα μέσον που υφίσταται θα πρέπει να αξιοποιείται για να μην σκουριάζει. Τι να πω, δεν θέλω να ασκήσω πολεμική, δηλαδή για ε, αναγάγεται, αναγάγεται το αυτό στα πυρηνικά, δεν πρέπει να σκουριάσουν και αυτά. Γιατί αυτό σημαίνει αυτό που λέτε, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μην σκουριάζουν. Είναι επικίνδυνη άποψη αυτή για να μην Σταματώ εδώ και νομίζω ότι ξεκαθάρισα αρκετά τις θέσεις μας. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθω σε μερικά από αυτά που υπόθηκαν. κυρία Κοπά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ για την σαφή και συνοπτική σας έκθεση. παρατήρησα πόσο απλή είναι σε σύγκριση με προηγούμενες πολυτεχνικές εκθέσεις που κάναμε. Πιστεύω ότι εμείς στις εκθέσεις μας πρέπει να χειριζόμαστε το θέμα της και είπαμε απλό και εύληπτο τρόπο για να το καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Φυσικά υποστηρίζω όλα όσα είπαν και οι σκιώδεις, ιδίως ο Γιάννης, αλλά υπενθυμίζω ότι η έκθεση επαναλαμβάνει πολλά από αυτά που ζητάμε εδώ και χρόνια. Η ενίσχυση, αυτονομία, λευκή βίβλο για την άμυνα και ασφάλεια, την οργάνωση των μάχημων ομάδων και παρόλα αυτά τα ζητάμε εδώ και χρόνια αλλά δεν έχουν γίνει πολλά. για αυτό το συμμερίζομαι τις επικρίσεις σας και τις θεωρώ σωστή βάση για συζήτηση. Η δυσκολία με την προώθηση της πρωτοβουλίας της Βαϊμέρης δείχνουν ότι δεν έχουμε ακόμη καταλάβει πώς ακριβώς θα γίνει το pooling και sharing. Τα εθνικά συμφέροντα υπερισχύουν ακόμη πρέπει να μπορέσουμε τελικά να είμαστε αποτελεσματικοί και οικονομικοί. Τις παραγράφους 51, 52 και 55 τις δέχομαι στη διατύπωσή τους, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι η δετερμινιστική γλώσσα της παραγράφου 50 δικαιολογείται. Μέχρι τώρα η, η αξιοπιστία της Ένωσης δεν έχει αμφισβητηθεί γιατί προέρχεται από πολλά παράγοντες και κυρίως από την νομοθετική και soft power που διαθέτει. Οι σοσιαλιστές δέχονται τις πρωτοβουλίες pooling και sharing ως μέσου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, αλλά ζητούν επίσης τη μείωση των αμυντικών προϋπολογισμών των χωρών μελών, ώστε τα ποσά που θα εξοικονομηθούν να διατεθούν για κοινωνικούς στόχους. Όσο για τις επιχειρήσεις, παρατήρησα πολλές επικρίσεις, άκουσα, και θα ήθελα να ξαναδούμε, να αποξιολογήσουμε εκ νέου τα αυτά τους αποτελέσματα, όπως το Χιούλεξ, Κόσοβο και άλλα που παρόλα αυτά νομίζω ότι έχουν θετική επίπτωση στη σταθεροποίηση της κατάστασης και βελτίωση των βιωτικού επιπέδων των βιωτικών του λαού εκεί. Τέλος, πολλά θα εξαρτηθούν από το κατά πόσον θα συμβουλευτούμε και άλλες σχετικές εκθέσεις την κυβερνοάμυνα, τη ρήτρα της αλληλεγγύης, τα κλιματολογικά θέματα και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ετήσια μα έκθεση για την ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πασκού τώρα. Well, thank you. Ευχαριστώ. Και πάλι η έκθεση είναι πολύ καλή όπως και η προηγούμενη και εκτιμώ ιδιαίτερα τις στρατηγικές συστάσεις, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μόνο γραφειοκρατική προσέγγιση χωρίς να σκεφτόμαστε που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη γενικότερη εικόνα. Οι στρατηγικές συστάσεις αυτές είναι καλές. Επίσης εκτιμώ το ότι ζητάτε λευκή βίβλο, διότι ξέρετε ότι υπήρξαν εκκλήσεις και πριν όταν ήταν ο προκάτοχός σας πρόεδρος. Ίσως ε, δεν είχε οριμάσει ο χρόνος, αλλά ίσως πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα είναι πώς θα βρούμε ισορροπία με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών. Τώρα, Μάλιστα καταγράφεται τις καινοτομίες στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, είναι τριών ετών ήδη. Σύντομα θα πάει στον υπηαγωγείο. Πρέπει λοιπόν να θυμίζουμε πάντοτε στον κόσμο και αν ας πούμε μιλήσουμε για την Τραπεζική Ένωση, η παρουσίαση των προϋπολογισμών στις Βρυξέλλες για αξιολόγηση Όλα αυτά δεν τα εφεύραν εκείνοι που υπέγραψαν τη συνθήκη της Λισαβόνας πριν από τρία χρόνια. Αυτοί απέχουν έτη φωτός. Αυτά τα πράγματα απέχουν έτη φωτός από τότε που υπογράφτηκε η συνθήκη της Λισαβόνας πριν από τρία χρόνια. Και όμως, ε, αρέσει η εκτίμηση των τωρινών επιχειρήσεων, τις ε, ικανότητες στρατιωτικές και πολιτικές. Ίσως το θέμα των εταιρικών σχέσεων μπορούμε να το επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο και ίσως να σκεφτείτε και ένα σημείο για την διατλαντική διασύνδεση, ιδιαίτερα τώρα που πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστον που πρέπει να διατηρήσουν οι ΙΠΑ. Τώρα που κοιτάζουν προς Ανατολάς. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για όλα αυτά που εκφράσατε και σαν εκτίμηση και τα σχόλια και τη βοήθειά σας. Τα σημείωσα όλα αυτά που είπατε θα εμπλουτίσουν την έκθεση. Κύριε Λέζιν, με ιδιαίτερη προσοχή άκουσα τις παρατηρήσεις σας να σας διευκρινίσω όμως δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, τα εργαλεία πώς χρησιμοποιούνται. Συμφωνώ. Δεν είμαι υπέρ της χρησιμοποίησής τους, όν και καλά, μια και υπάρχουν ε, και κάτω οποιασδήποτε συνθήκες. Και να σα ε, υπενθυμίσω ότι τα πυρηνικά όπλα όπως ε, τα έχουμε συλλάβει εμείς είναι αποτροπής και αποθάρρυσης και όχι χρήσης λοιπόν ε, μια και υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα, να τα χρησιμοποιήσουμε κιόλας όχι, δεν τίθεται, δεν έχει τεθεί ποτέ έτσι το θέμα. Δεν είμαι σόν και καλά επίση ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία επειδή υπάρχουν αλλά στην ΚΥΠΑ και στην κοινή πολιτική ασφάλειας άμυνας όλα αυτά ε, έτσι ε, πραγματιστικά φτιάχτηκαν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Ε, η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας ε, αυτή και οι ενέργειες λόγω των κρίσεων παντού και στα Βαλκάνια ας πούμε ε, καταβλήκαν προσπάθειες όπως και από τον Χαβιέ Σολανά και μάλιστα με τρόπο όχι καθόλου αφηρημένο ή δογματικό. Το ίδιο ισχύει και σήμερα και ορισμένα εργαλεία όταν λέω ότι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν, το λέω επειδή θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε στιγμές κρίσης έτσι και με τα μέσα που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε, θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ας πούμε στην περίπτωση της κρίσης στη Λιβύη χωρίς όμως οπωσδήποτε μια στρατιωτική παρέμβαση από λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέραμε και σήμερα ότι και διπλωματικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους θα ήταν εντελώς αδύνατοι. Εντάξει, Επαναλαμβάνω, δεν είμαι υπέρ τη υποχρεωτική χρήση των όσων υπάρχουν μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν, αλλά μερικέ φορέ μπορεί πραγματικά να μα χρησιμεύσουν για τα οικονομικά συμφέροντα. Ναι, ακούσαμε την ερώτηση αυτή. Δεν είναι ότι θα πρέπει την πολιτική να την επιδιώξουμε για ε, να πετύχουμε στόχους οικονομικούς μέσω στρατιωτικών ενεργειών. Εδώ τα κράτη ομέλη όμως έτσι κι αλλιώς έχουν μια βιομηχανία σημαντική για αμυντικούς σκοπούς ε, με πλατιά παραγωγή, όχι στενά αυστηρά στρατιωτική και η παραγωγή αυτή δημιουργεί θέσεις απασχόλησης αλλά και καινοτομία, πλούτο τεχνολογικό. Άρα λοιπόν επικίνδυνο θα ήταν σε αυτό το σημερινό κόσμο τα κράτη μέσα Ευρωπαϊκή Ένωσης να μην έχουν αυτές τις γνώσεις τις βιομηχανικές και να τις χρησιμοποιούν. Και το δεύτερο μέρος, τις σχέσεις με τη βιομηχανία. Να σας πω ότι πάει προς την βιομηχανική πτυχή. Όχι, δεν θα πρέπει να το φοβόμαστε και να το λέμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γνωρίζει πώς θα υπερσπίζεται τα συμφέροντά της και τα εμπορικά, όπως ας πούμε κατά των πειρατών ε, στα ανοιχτά της Σομαλίας και αυτό έχει μια διάσταση προστασίας των εμπορικών συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τα πλοία τα δικά μας, ο στόλος ο δικός μας έχουν το 30% του εμπορίου στην περιοχή αυτή και υπάρχει μια σοβαρή απειλή λοιπόν στην Ευρώπη, όχι μόνο στο εμπόριο αλλά και στην ίδια την Ευρώπη. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τα μέσα στα χέρια της για να αντιμετωπίσει παρόμοιες απειλές. Εντάξει, σίγουρα όμως θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αυτή και οι πολιτικές ομάδες άλλωστε θα αποφασίσουν πάνω στο τι θα θέλουν να ακολουθήσουν σαν προσανατολισμούς. Μάικελ, μόλις ήρθε. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Ήμουν στην Επιτροπή Μεταφορών και μιλήσαμε για το πακέτο των αεροδρομίων. Γι' αυτό δεν μπορούσα να έρθω και εδώ. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρό μας για το σχέδιο έκθεσης. Ε, συμμερίζομαι όλες τις πολιτικές του εκτιμήσεις. Νομίζω ότι είναι και μια συνεκτική προσέγγιση, comprehensive approach, όπως λέμε, για την πολιτική μας σε αυτό το τομέα και όλα όσα έπρεπε να υποθούν, τα Θα κάνω κάποιες ε, προσθήκες εκεί όπου σε προηγούμενες εκθέσεις είχαμε ασκήσει συγκεκριμένη κριτική στο Συμβούλιο σχετικά με όσα δεν έγιναν, δηλαδή αναφερόμενοι στις προτάσεις μας που δεν ε, υλοποιήθηκαν, για να εμπλουτίσω λίγο την έκθεση πιστεύω. Άλλωστε είναι ε, καθήκον μας και ε, απέναντι στα, να ασκήσουμε πιέσεις και ε, στα κρατημέλη και στην κυρία Άστον σχετικά με το τι πρέπει να, να κάνει η πολιτική εν ώψη των διεθνών εξελίξεων. Θα πρέπει να προχωρούν στην, τάξη και, στην πράξη. Και σε αυτό αυτό το τομέα της πολιτικής μόνο από κοινού μπορούμε να επιτύχουμε πράγματα, διότι με μονομένα κράτη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις προκλήσεις και στις απειλές που γίνονται όλο και πιο μεγάλες. Και ε, εν ώψη μιας δυνητικής ε, απόσυρσης του, των συμμάχων μας ε, από αυτή την περιοχή πρέπει και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε και να αναπτύξουμε αυτό αυτόνομες ικανότητες προς το συμφέρον των πολιτών μας και στην εσωτερική και στην εξωτερική ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να δώσουμε τέτοιες οικονομικές επίσης εγγύσεις. Τέτοιου είδους ε, διευκρινήσεις θα κάνω στην έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και αν κάποιος άλλος δεν θα επιθυμεί να λάβει το λόγο, θα περιοριστούμε σε αυτά στη σχετική συζήτηση και να δούμε μετά από τη κατάσταση τροπολογιών το μεσημέρι 21 Σεπτεμβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες και 9 Οκτωβρίου θα τα πούμε και πάλι όπως και με την έκθεση Πασκού για νέα συζήτηση. Βέβαια θα συναντηθώ με τους ε, μέχρι τότε, με τους κοιόντες συγκητές. Σας ευχαριστώ. Αυτά. Κλείνει η συνεδρίαση. Το Προεδρείο θα συνεδριάσει τάχιστα για 10 λεπτά. Ευχαριστώ.